Herr Präsident! Bitte nehmen Sie. Ich erkläre die am 3. April unterbrochene Sitzung. Κυρίσω την επανάληψη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε διακοπεί στις 3 Απριλίου. Κυρίες και